Συνεχίζουμε συνεδρία της Ολομέλειας με τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της κυρίας Τσιούτε και θα απαντήσει ο κύριος Ζόναρ. Τι ε, Violence against women constitutes a violation of η βία κατά των γυναικών είναι παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι δεσμευμένη στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων της. Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με τα ήθη και έθιμα ούτε από θρησκευτικές παραδόσεις. Επαναλαμβάνει λοιπόν η Κομισιόν τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, πράγμα που φαίνεται και από τη δήλωση του Απριλίου 2010 για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που τονίζει ιδιαίτερα την προστασία των θυμάτων, εγκλημάτων ο, μεταξύ των οποίων και η βία κατά των γυναικών και, η, και ο σεξουαλικός ακροτηριασμός. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε μία άλλη στρατηγική καινούργια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και πρόκειται στο πρώτο ήμιση του 2011 να εγκρίνουμε τη στρατηγική αυτή καταπολέμησης της βίας επαναλαμβάνω κατά τον γυναικών. Το περασμένο Μάρτιο ενδυναμώσαμε τη γενική μας δέσμευση για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ας το πω. Όπως συζητήθηκε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουνίου, η χάρτα αυτή προτείνει την εφαρμογή ενός συντονισμένου πλαισίου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και ενδυνάμωση της δράσης μας και με νομοθετικά και με άλλα μέσα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ σήμερα ανακοίνωσε μία στρατηγική για την ισότητα των φύλων και ένα συνολικό σχέδιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Η βία κατά των γυναικών είναι ουσιώδες τμήμα επαναλαμβάνουμε και θα προστατεύσουμε τα θύματα κατά της βίας αυτής. Η Κομισιόν εγκρίνει με τα χαράς το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την βία κατά των γυναικών και την κατάργηση της βίας αυτής κατά των γυναικών γυναικών γιατί θέλουμε να αποτραπεί η βία κατά των γυναικών. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μελέτη αξιολόγησης για να δούμε ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες νομοθέτησης για την καταπολέμηση της βίας και κατά των γυναικών και κατά των παιδών. Και τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής θα παρουσιαστούν στην ε, διάσκεψη υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2010. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ και τώρα οι δύο συμπληρωματικέ μαζί. Πρώτον κυρία Λίνκοβιτς Γιούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εκτενή απάντησή σας. Θα ήθελα πάντως ε, να σας επισημάνω ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά συγκρίσιμα στοιχεία, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε δείκτες για τη βία κατά των γυναικών. Προτιθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για εθνικά σχέδια δράση για συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων προκειμένου να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν δεν έχουμε σαφή γνώση για την κατάσταση, δεν μπορούμε να προτείνουμε και κάποιες αλλαγές. Yeah, thank you. Uh, aus Angst äh, verschweigen Λόγω του φόβου οι γυναίκες ε, πολλές φορές ε, κρύβουν την άσκηση βία εις βάρος τους ε, στο, στα σπίτια τους. Αυτό είναι γνωστό από την Amnesty International. Στην Τουρκία μέχρι το 50% των γυναικών δέχονται σωματική βία στις οικογένειές τους. Και τίθεται το εξής ερώτημα. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπόνηση αυτής της μελέτης κατέστη άραγε δυνατό να ερευνηθούν και οι περιπτώσεις στην Τουρκία Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Επίτροπος. Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως ότι είναι πολύ σημαντική η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και για τη δημιουργία δικτών. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η συλλογή στοιχείων και η ανάπτυξη των καταλήλων δικτών θα γίνει, θα είναι τμήμα της στρατηγικής την οποία ανέφερα προηγουμένως. Επίσης μπορώ να σας διαβεβαιώσω κύριε βουλευτέ ότι το θέμα θα το θέσουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Την καταπολέμηση δηλαδή κατά των γυναικών ιδιαίτερα στις χώρες που βρίσκονται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις και που, διότι έχουμε πολύ τακτικές επαφές και δυνατότητα να συλλέξουμε τα στοιχεία αυτά όπως πρέπει. Ευχαριστούμε, Επιτροπέ, πάρα πολύ. Περνάμε στην ερώτηση της κυρίας Χάρκιν τώρα για τον κανονισμό 1083, ερώτηση υπερθυμών 22. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για την ερώτησή της όπως ξέρετε, τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως το Αναπτυξιακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο, υπόκεινται σε μεικτή διαχείριση. Η διαχειριστική αρχή που έχει καθοριστεί από τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων. Επίσης, ε, εξασφαλίζεται η σωστή επιλογή ε, των προγραμμάτων για τη συγχρηματοδότηση ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν ε, στα κράτη-μέλη και με βάση και τους κοινωτικούς κανονισμούς. Υπάρχουν δύο μνήες ό,τι αφορά την ανακατανομή στον Γενικό Κανονισμό 1083 του 2006 που προβλέπει τις γενικές διατάξεις για το Περιφερειακό Ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Στο ιδεολογική σκέψη 42 προβλέπεται ότι σε ό,τι αφορά τα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, τα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει όλε τι απαραίτητες πληροφορίε, προκειμένου να ε, εξασφαλίσει ότι η συνεισφορά από το Διαρθρωτικό Ταμείο δεν θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων απασχόληση οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υποστηρίξει κοινωτική χρηματοδότηση με την κατάσταση μια επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το άρθρο 47 προβλέπει ότι οι διαχειριστικέ αρχέ των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συγχρηματοδοτούμενε επενδύσει ε, διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση ε, μια επιχείρηση. Όταν μια εταιρεία δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, ε, γίνεται ανάκτηση της κοινωτικής συνεισφοράς. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση, ένα πρόγραμμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τις επενδύσεις αυτών των άρθρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να ενημερώσει σχετικά τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε επιχειρήσεις που είναι ε, το αντικείμενο μιας διαδικασίας ανάκτησης δεν θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά κονδύλια για τις δραστηριότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται για διαχείριση των τέτοιων δραστηριοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Βιωτικών Συνθηκών. Σε περίπτωση κρατικών ε, προγραμμάτων, και εκεί υπάρχει απέτηση, να διατηρηθεί απέτηση για μια πενταετία, για τις περιφερειακές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις απασχόλησης. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ένα χειρίδιο που προβλέπει και τις δυνατότητες ε, ε, ενημέρωση για τις εξαιρέσεις και τις μαζικές, ε, τις συλλογικές εξαιρέσεις. Επαναλαμβάνω, οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να εκδίδουν και κατάλογο δικαιούχων των διαφόρων συνεισφορών και των ποσών που δικαιούνται επίσης. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και στο σελίδα των, του Κοινωνικού Ταμείου και αντίστοιχε ιστοσελίδε των διευθυντικών ταμείων υπάρχουν και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν, συμπληρωματική. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την διεξοδική του απάντηση. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μία συνέπεια της βιομηχανικής μας πολιτικής και μία συνοχή. Αναφερθήκατε στην αιτιολογική σκέψη 42 και Είπατε ότι η κοινωτική χρηματοδότηση δεν θα υποστηρίξει με την κατάσταση και ότι οι χρηματοδοτούμενε επενδύσει θα πρέπει να διατηρούνται για μία πενταετία. Τι γίνεται όμω μετά τη χορήγηση τη ε, χρηματοδότηση, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι μία εταιρεία δεν θα πωλήσει πουθενά στη, στα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη εργαζόμενους. Μπορούμε να ελέγξουμε ή να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και αν όντω ε, λάβει χώρα τέτοια πώληση σε άλλο κράτος μέλος, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χάρκιν, υπάρχει μηχανισμός ε, τέτοιας παρακολούθησης και μάλιστα το Κοινωνικό Ταμείο έχει γραφεί σε όλα τα κράτη-μέλη και έχει στενές σχέσεις με τις διαχειριστικές αρχές. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης της κατάστασης ε, σε πολλά κρατημέλη ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και αν ε, γίνουν τέτοιε απολύσεις, υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών και εν ανάγκη και εφαρμογής διορθωτικών μέτρων. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν βλέπω τον κύριο Σεκέρσκι στην αίθουσα. Οπότε η ερώτησή του καταπίπτει. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις που δώσατε και για την παρουσία σας φυσικά. Θα ζητήσουμε τώρα από τον κύριο Έτιγκερ να έρθει στο βήμα. And the first question to Mr. Η πρώτη ερώτηση για τον κύριο Έτιγκερ είναι η ερώτηση παριθμών 24 του κύριου Ταραμπέλα. Όποτε είστε έτοιμο κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Βλέποντα τι τιμέ ενέργεια Βλέποντας τις ε, τιμές ενέργειας ε, και γενικότερα ε, την αύξηση αυτών ε, τον τελευταίο καιρό και αν ε, αναλύσουμε την αύξηση των τιμών καταλήγουμε σε διάφορα συμπεράσματα. Η Κομισιόν λοιπόν έλαβε μία σειρά μέτρων και στις περιπτώσεις των γερμανικών επιχειρήσεων και στην περίπτωση της σουηδικής επιχείρησης. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν τις ε, τιμές ενέργειας ε, στην Ευρώπη. Στις ε, αρχές του μήνα τόνισα στους Υπουργούς Ενέργειας ότι οι διατάξεις για την εσωτερική αγορά ενέργειας έχουν την προστασία του καταναλωτή ως απόλυτο στόχο. Θέλουμε λοιπόν, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ορίσουμε με σαφήνεια τις τιμές, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και όσον αφορά τις, ε, ε τους λογαριασμούς ε, που στέλνουν τους καταναλωτές, εκεί ε, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον, την δομή των λογαριασμών. Ο στόχος λοιπόν είναι να υπάρχουν, υπάρχει ανταλλαγή πρακτικών, ένα σωστό benchmarking και κατόπιν τούτου, κάτω από το πρίσμα συζητείται ε, το θέμα της ενέργειας. Εμείς έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει το θέμα και η, έρευνα, η μελέτη που έχει ε, εκπονηθεί είναι ε, προσπελάσιμη σε όλους. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο περιλαμβάνει και νέες διατάξεις για το πόσο συχνά θα γίνεται η καταμέτρηση της ενέργειας και για την σωστή κατανάλωση. Όλα αυτά θέλουμε να τα προάγουμε. Και υπάρχει ένας χάρτης ε, για τη σωστή κατανάλωση ενέργειας, ένας χάρτης ε, που ε, δημοσιεύθηκε πριν από τρία χρόνια. Σε πάρα πολλές οδηγίες και σε πάρα πολλά εθνικά εφαρμοστικά μέτρα αναφέρονται διάφοροι κανονισμοί δεσμευτικής φύσεως. Το θέμα αυτό λοιπόν θα το εξακολουθήσουμε να το επεξεργόμαστε από κοινού τους Υπουργούς Ενέργειας. 8.30 θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε. Οπότε θα ακούσουμε τις ε, απαντήσεις σε ερωτήσεις του Ταραμπέλα, Τικάου, Χουντή και Γιακολίνο, αλλά δεν νομίζω θα προλάβουμε να ακούσουμε απαντήσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Ταραμπέλα και μετά η κυρία Τιτσάου. Ευχαριστώ. Μία ε, έκθεση Τη Εθνική Τράπεζας του Βελγίου δείχνει πόσο ρευστές είναι οι τιμές ηλεκτρισμού αλλά και τι προβλήματα υπάρχουν για τον καταναλωτή. Πολλαπλά είναι τα προβλήματα που ανέκυψαν με τους παραγωγούς μετά την απελευθέρωση και μάλιστα ο Ομοσπονδιακός ε, Ρυθμιστής στο Βέλγιο, η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή είπε ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην αγορά και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση του καταναλωτή του καταναλωτή ενέργειας δεν θα πρέπει η απελευθέρωση να γίνει ξέφραγο αμπέλι ε, και να αφήσει ελεύθερους τους παρόχους ε, για να κάνουν κατάχρηση των εξουσιών τους. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να καταρτήσουμε μια πραγματική χάρτα των καταναλωτών. Η κυρία Τσικάου για μισό λεπτό. Thank you, Mr. Chair, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για να, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες που αφορούν την κατανάλωση των οικοκυριών της Ευρώπης, θα έπρεπε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο γενικότερο πλαίσιο, κάποια μήνυμο πληροφόρηση που πρέπει να εμφαίνεται στα τιμολόγια για να μπορούν οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες να το καταλαβαίνουν. Κύριος Μάγκερ, 30 δευτερόλεπτα. Το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, αυτό είναι διαμφισβήτητο, γιατί χωρίς ε, διαφάνεια δεν υπάρχει υγιή ανταγωνισμό ε, και χωρίς υγιή ανταγωνισμό δεν υπάρχουν και ικανοποιημένοι καταναλωτές. Μόνο που ερωτώ το εξή ε, έχουμε κάποιους παρόχους που αρνούνται να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του, και αυτό το κάνουν για να εμποδίσουν άλλους να εισέλθουν στην αγορά. Εδώ η Κομισιόν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και αν ναι, με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις πολύ σωστά τέθησαν και καταδεικνύουν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ε, έχει νόημα μόνο εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός, διαφάνεια και η δυνατότητα μεταφοράς από το χώρο παραγωγής στο χώρο της ε, κατανάλωσης. Εμείς με το πακέτο μας ε, περί κοινή αγοράς είμαστε στο σωστό δρόμο και πολλές ε, διατάξεις ε, και πολλές ε, καταγγελίες που έχουν γίνει δείχνουν στα κρατημέλη που έχουν προβεί σε παραβιάσεις. Ελπίζουμε το δεύτερο πακέτο σύντομα να το έχουμε στα χέρια μας. Για το τρίτο θα περιμένουμε μέχρι την επόμενη άνοιξη και μέχρι τότε όλοι θα πρέπει να θεωρούν και να περιμένουν να δουν τι θα έχει γίνει με την ολοκλήρωση. Κάποια δίκτυα που υπάρχουν παρότι υπάρχει ζήτηση δεν τη χάνουν πλήρους εκμετάλλευσης. Αν εσείς έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί εμείς ερευνούμε αυτές τις ε, περιπτώσεις, καθότι ο στόχος μας είναι για όλους να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας και με τους ίδιους όρους. Αυτό ισχύει και για το αέριο, όπου πράγματι εκεί υπάρχει ε, κάποια έλλειψη δικτύων. Κατά τα άλλα, στις αρχές του έτους ε, θα δημοσιεύσουμε και μία ενδιάμεση έκθεση για την κοινή αγορά, να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, ε, το κοινοβούλιο, αλλά και η πολιτική, η εθνική πολιτική να γνωρίζουν ε, τι γίνεται ας πούμε με το θέμα του αερίου. Γιατί για το αέριο πολλοί εκφράζουν ε, πανηγυρικούς αλλά στην, πρακτική, στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Τώρα, όσον αφορά την διαφάνεια στις ε, καταμετρήσεις και στους λογαριασμούς, και εμείς αυτό επιθυμούμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη που εφαρμόζουν Τη διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ νομίζω ότι παράλληλα με την κοινή αγορά πρέπει να προβληθεί και το θέμα της εκπαίδευσης του καταναλωτή. Είναι δύο θέματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα θέματα αυτά απαιτούν ε, επαγρύπνηση στον προϋπολογισμό, απαιτούν ε, τις ε, αρμοδιότητες αλλά και τον ανταγωνισμό. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες για να καλύπτονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στην κοινή αγορά. Ευχαριστούμε. Και τώρα η ερώτηση 25 της κυρίας Τικάου για θέματα περιφερειακής συνεργασίας στην ενέργεια. Όταν ο Επίτροπος είναι έτοιμος μπορεί και να μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, αυτό που σας ενδιαφέρει, το να υπάρχει μια ευφυής υποδομή ε, ενέργειας, εμείς αυτό το χαιρετίζουμε. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που υπάρχουν τα ερμηνεύουμε πολύ προσεκτικά. Έχουμε μία έρευνα της Κομισιόν ε, πριν από δύο χρόνια που κατέληξε στο ότι η πρωτογενής ε, κατανάλωση ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειωθεί κατά 9% και με βάση τις μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος θα προκύψει μια σημαντική εξοικονόμηση. Βλέπουμε λοιπόν αυτό προκύπτει, μάλλον θα ωφελήσει και την τεχνολογία και την ασφάλεια και την αγορά και τον καταναλωτή. Ε, θα μπορούμε να έχουμε ευφύ έλεγχο, καλύτερη διαχείριση και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα πλεονεκτήματα δεν μπορεί βέβαια να τα έχει κανείς ε, δωρεάν, γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις. Ορισμένα κράτη-μέλη έκαναν τα πρώτα βήματα για την εγκατάσταση των δικτύων. Σουηδία, Ιταλία, ε, περίπου το 100% των ε, πελατών τους το έχουν εξοπλίσει με ευφυή e συστήματα καταμέτρησης. Προγράμματα υπάρχουν στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Η Κομισιόν λοιπόν προάγει, στηρίζει αυτή την υποδομή του να υπάρχουν ευφύ e συστήματα καταμέτρησης και τα σχετικά δίκτυα. Ε, υπάρχει η οδηγία που έχει εκπονηθεί από αυτού. Συστήσαμε επίσης και μία ομάδα εργασίας μια ε, ομάδα εργασία που ασχολείται συμφέροντα της βιομηχανίας ε, και των καταναλωτών. Εξετάζονται ε, τα κίνητρα, η σκοπιμότητα, προσπαθεί να εντοπιστεί που υπάρχουν ανάγκες, την τεχνολογία και την επόμενη χρονιά θα έχουμε το αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας και θα το παρουσιάσουμε επίσημα εδώ στο Κοινοβούλιο. Mm. Τώρα, όσον αφορά την ανακοίνωση ε, που αφορά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Αυτή η ανακοίνωση έχει πολλούς στόχους και δεν αφορά μόνο την ευφύη καταμέτρηση. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται στο να συμπεριληφθούν ε, τα κράτη-μέλη στις διαβουλεύσεις ε, για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και περιφερειακών διασυνδέσεων θέλουμε να καλύπτουμε πολλές μεγάλες περιοχές και να μπορούμε να κάνουμε και έναν απολογισμό. Εδώ βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον οργανισμό για την συνεργασία, την ΕΖΑ. Πρέπει να προβάλλουμε το ρόλο αυτού του οργανισμού που θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του επόμενου έτους. Επιθυμούμε λοιπόν τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και μέσω της ε, περιφερειακής ε, συνεργασίας τους ε, στόχους αυτούς να τους προβάλλουμε. Η κυρία Τικάο. Μισάρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κύριε Επιτρόπε να σας ρωτήσω ακόμη κάτι γιατί τα smart grids, αυτά τα ευφύ δικτύα, θα συμβάλλουν τα μάλα στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ή όπου ε, υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές. Προβλέπονται κάποιες επενδύσεις μέσω και μακροπρόθεσμα και στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Κύριε ναι. Πίτρο, έχετε το λόγο.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 θα προλάβουμε να ακούσουμε και την απάντηση του κύριου Γιακολίνο, αλλά οι υπόλοιπε ερωτήσει 28-30 θα απαντηθούν δυστυχώ γραπτώ. 28-32. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την ερώτηση 26. Sie sprechen den griechischen Energiesektor an. Εσείς στον ε, ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και στην αναδιάρθρωσή του μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει ότι με το άνοιγμα της αγοράς για τον ανταγωνισμό ε, θα γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων και με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ανάπτυξη και θέση εργασία στον ενεργειακό τομέα. Και αυτά θα επιδράσουν θετικά και σε άλλους ε, τομείς της οικονομίας εναπόκειται στην Ελλάδα να αποφασίσει πώς θα αναπτύξει τον ενεργειακό της τομέα, πώς θα δημιουργήσει νέες δομές το unbundling, δηλαδή το καθεστώς ιδιοκτησίας ε, στο δίκτυο ε, διανομής ε, ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για να προάγει κανείς τον ανταγωνισμό. Και ως έχει κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι δημοσιονομικής φύσεως για την Ελλάδα να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει και για τον την εκποίηση ε, ενός τμήματος ε, των λιγνητικών και υδρολεκτρικών μονάδων της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, γιατί σας λέω πρόκειται για έσοδα και ανταγωνισμού. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ελληνικού κράτους να αποφασίσει το τι θα κάνει. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η ΔΕΗ ως ε, μόνος πάροχος αυτή τη στιγμή να μπορέσει να υποφεληθεί από τα ε, θετικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθυστέρηση στην Ελλάδα ε, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της ε, ε, και πρέπει να επιταχύνει σε θέματα ανταγωνισμού. Εμείς είμαστε σε καλό διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση και αυτό είναι σημαντικό. Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολύ εντυπωσιακά μέτρα στον τομέα των δημοσιονομικών και γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση στην Ελλάδα η συνεργασία αυτή βασίζεται πάνω στην εταιρική σχέση. Όσον αφορά τις τιμές ε, καταναλωτή. Η ε, κυβέρνηση έχει ορίσει κάποιες κατηγορίες, ε, αυτές όμως οι κατηγορίες δεν είναι ενιαίες και σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση εξορθολογισμού των τιμολογίων και η δική μας ε, η άποψη ότι το, οι τιμές θα πρέπει να ορίζονται με βάση το κόστος να είναι ένα κίνητρο για τον καταναλωτή να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας και για τις επιχειρήσεις κίνητρο για να κάνουν επενδύσεις. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρκετά χαμηλές και διότι υπάρχει ε, παραγωγή ε, λιγνίτη, έχουμε υδρολεκτική ενέργεια. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μεγάλες Ε, Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει βέβαια και μείωση της ζήτησης. Κατά τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν άλλοι παράγοντες, δηλαδή όλο και μεγαλύτερη χρήση αερίου που είναι ακριβό αυξανόμενο περιβαλλοντικό κόστο, και οι τιμέ στην Ελλάδα θα αυξηθούν Επίσης θα μειωθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια γιατί πλέον δεν έχουμε μεγάλες βροχοπτώσεις, είναι σε φυσιολογικό ρυθμό. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές ε, και αυτή η αύξηση των τιμών ε, είναι άσχετη με την απελευθέρωση της αγοράς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το σύστημα να είναι όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται και οι αυξήσει των τιμών να παραμείνουν όσο το δυνατόν σε χαμηλότερο επίπεδο, πράγμα που θα είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ο κύριος Χατζηγεωργίου πρώτα, μετά η κυρία Ποδηματά και μετά ο κύριος Παπενικολάου για συμπληρωματικές. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Κύριε Επίτροπε, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο τη Ελλάδα, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια τη ηλεκτρική ενέργεια αντανακλούν σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 τι τιμέ χονδρικής τη αγορά δηλαδή ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει την τιμή του ρεύματο ει βάρο των καταναλωτών και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων και τη οικονομία. τι επιπτώσει θα έχουν αυτά τα μέτρα στην παραγωγή και την ανάπτυξη τη ελλάδα με αυτά τα μέτρα δηλαδή με αυξήσει τιμολογίων θα βγει η ελλάδα από την κρίση και την κυδαιμονία του διεθνού νομισματικού ταμείου? και τέλο μόλι την περασμένη εβδομάδα πήραμε απάντηση από τον κύριο ρεν για την έκρηξη στον πληθωρισμό που φτάνει στο 5,6 τι επιπτώσεις θα έχουν τα παραπάνω μέτρα στον πληθωρισμό. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Thank you, Mr. Podimata. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην απάντησή σας στο διαχωρισμό των συστημάτων μεταφοράς θέλω να σας ε, ζητήσω αν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι η ελλάδα όπως και όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης είναι ελεύθερα με βάση το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας 72 του 2009 να επιλέξουν ένα από τα τρία ισοδύναμα μοντέλα για το διαχωρισμό του συστήματος μεταφοράς και ότι δεν είναι θέμα της επιτροπής να υποδείξει στα κράτη μέλη ποιο από τα τρία μοντέλα θα αποφασίσουν να υιοθετήσουν. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ΔΕΗ είναι μια κερδοφόρα και σχετικά υγιής επιχείρηση παρά την σημαντική πτώση των κερδών της τη φετινή χρονιά η οποία κυρίως οφείλεται στην οικονομική κρίση και την μειωμένη κατανάλωση. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Πριν προχωρήσει σε αυτές τις προτάσεις η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε μελέτες για τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια πρόταση σε ό,τι αφορά τη θέση της εταιρείας στην αγορά της ενέργειας σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση και την κερδοφορία της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ τι εξελίξει στην Ελλάδα με μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό. Σεβασμό απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία εν ώψη της κατάστασης, με την κατάσταση που ισχύει, έχει το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Έχει λάβει μέτρα, εξοικονομήσει, ε, μεταρρυθμίσει και η κυβέρνηση αυτή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ευρωπαϊκούς φορείς και με άλλους παγκόσμιους φορείς δεν φίδεται προσπαθειών για να σταθεροποιήσει τον προϋπολογισμό, τα δημοσιονομικά και να συμβάλλει στη σταθεροποίηση του ευρώ. Βεβαίως ε, δεν πρέπει να χάνουμε το σύνολο, το πλαίσιο. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα μορατόριο. Δεν μπορούμε να αναστείλουμε τους κανόνες της αγοράς. Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο δικαιωμά μου, αλλά υποχρέωσή μου να οθήσω τις εξελίξεις ε, προς την ε, απελευθέρωση των κανόνων της αγοράς, ε, την κατάργηση μονοπωλίων, να έχουμε ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Οι κανόνες της αγοράς είναι πολύ παλαιότεροι από την παρουσία μου στην Κομισιόν και το unbundling είναι ενός έτους, περίπου όσο και εγώ στην παρουσία μου στην Κομισιόν. Εγώ λοιπόν είμαι πρόθυμος αυτό το μνημόνιο συναντήληψης να μην το ερμηνεύω ερμηνεύω περιοριστικά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Παραδείγματος χάνει το unbundling, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός. Δεν μου επιβάλλει να πουληθούν τα δίκτυα. Εμείς ε, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ο μέχρι τώρα ιδιοκτήτης που δραστηριοποιείται στην ενέργεια να μην ασχολείται με και να μην παρεμβαίνει στις λειτουργικές ενέργειες της θηγατρικής εταιρείας, το δίκτυο να είναι ανοιχτό σε όλους όσοι επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι να μπορούν να εμφανιστούν και ανταγωνιστές για το αέριο και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Κομισιόν προσπαθεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα δημοσιονομικά αλλά και για τα συμφέροντα της Ελλάδας στην ενεργειακή αγορά. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στην ερώτηση 27 του κυρίου Γιακολίνο. Αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση προς το συγκεκριμένο επίτροπο και αφορά τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Παριθμόν 27 ερώτηση κύριε επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα είναι ε, πρώτης προτεραιότητας ε, στα θέματα που με ενδιαφέρουν. Εδώ στην Ολομέλεια μιλήσαμε ε, έτσι ώστε στην Ευρώπη και σε γειτονικές περιοχές να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ποια είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα και θέλουμε να διασφαλίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν ε, οι βέλτιστες ε, δυνατές προδιαγραφές και αυτό προϋποθέτει στενή συνεργασία ε, με τις ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνεργασία με τις αρχές οι οποίες κάνουν και τις επιθεωρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη στις offshore δραστηριότητες να εφαρμόζουν τους ίδιους ενιαίους αυστηρούς ελέγχους. Επίσης, όσον αφορά την έγκριση των δραστηριοτήτων offshore ε, με βάση το ισχύον δίκαιο, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, εγώ λοιπόν όσον αφορά τις offshore δραστηριότητες ε, θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει κάποια αναστολή των ε, αδειών, ε, κυρίως όταν υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις. Ορισμένα κρατημέλη, κυρίως η Ιταλία, αποφάσισαν ένα τέτοιο, να ακολουθήσουν ένα τέτοιο προληπτικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Και καταρχήν ε, πρόκειται για ευρωπαϊκές περιοχές, ε, για τη Μεσόγειο. Έχουμε λοιπόν κοινά συμφέροντα στον περιβαλλοντικό τομέα, γιατί αν γίνει ατύχημα στα ε, ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτομάτως θα υπάρχουν επιπτώσεις σε μεγαλύτερες περιοχές και τα Νάπαλιν. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία στην Αλγερία και στη Λιβύη. Και η οι υπουργοί ε, πρότειναν συνεργασία και το ε, Υπουργείο ακολουθεί λοιπόν το στόχο να προτείνει υψηλές ε, προδιαγραφές περιβάλλοντος. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, έχουμε ε, εισαγάγει αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές. Οι ευρωπαϊκές νομικές διατάξεις νομίζω ότι πρέπει να περιβάλλουν ενιαίες διατάξεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξουν και μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις δηλαδή να ισχύει το περιβαλλοντικό δίκαιο έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των ε, επιπτώσεων. Και στο τέλος αυτού του έτους ε, θα έχουμε την τελική μελέτη. Εάν υπάρξουν, εάν μπορούμε να καταθέσουμε καλύτερες ε, προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές ποινικέ διώξεις. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ε, και πρόληψη και ασφάλεια αλλά και έκτακτα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τα χωρικά ύδατα των ε, γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες που έχουν αυτές οι χώρες απέναντι σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιστάσεις και επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι η χρηματοοικονομική επιφάνεια αυτών των επιχειρήσεων και οι δυνατότητές τους. Γιατί οι επιχειρήσεις αυτές και οι εταιρείε θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλουν αποζημιώσεις σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν, να επαληθεύσουμε το κατά πόσο οι εταιρείε αυτέ είναι δεόντω ασφαλισμένε, ώστε να μπορέσουν να καταβάλουν τι αποζημιώσει σε περίπτωση καταστροφή. Έτσι μόνο θα εγγυηθούμε το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και για τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά και για το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και περιμένουμε ε, δελεχή συζήτηση στην Αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ο κύριος Γιακολίνο, μετά ο κύριος Ρούμπιχ και μετά η κυρία Μορκουνάιτε Μικουλέιρινε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δώσατε χρόνο Ευχαριστώ επίσης και τον Επίτροπο. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Φυσικά η εγγύηση που προσφέρει ο Επίτροπος ε, είναι πολύ θετικές. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει δυνατότητα επέμβασης ε, ή μάλλον διαβήματος προς τις ε, αρχές της Λιβύης ώστε όντως να λάβει χώρα αυτό το μορατόριο ώστε να υπάρξει συντονισμός για τη Μεσογειακή Λεκάνη και να υλοποιηθεί το σχετικό σχέδιο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σουρουμπίχ. Äh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ποια διεθνή εργαλεία διαθέτουμε για να επιβληθεί κάποια τάξη εδώ στον διεθνή ανταγωνισμό έτσι ώστε όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες αλλά και να αναλαμβάνουν το ίδιο κόστος σε περίπτωση ανάληψης κινδύνου διότι αλλιώς μπορεί να μην έχουμε τις απαραίτητες δομές και οι διαδικασίες αδειοδότηση είναι τόσο αργές που μπορεί να βρεθούμε καθυστερημένοι. Δεν μπορώ να προφέρω το όνομά σας σωστά, αλλά εννοώ ότι δεν μπορούμε το ερώτημά σας κυρία Μορκουνάιτε Μικουλενιένε να το χειριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως δεν θα έχω το χρόνο να θέσω το συμπληρωματικό μου ερώτημα, αλλά και αυτό που συζητήσαμε πριν με ενδιαφέρει. Πρέπει να ενδυναμωθεί το νομοθετικό σύστημα που αφορά το περιβάλλον και τις πετρελαϊκές γεατρήσεις. Ποια κατάσταση λοιπόν ισχύει στη Μεσόγειο είναι γνωστή, αλλά εγώ ερωτώ κάτι για τη Βαλτική, διότι γνωρίζω, γνωρίζω ότι πρέπει με να λάβουμε υπόψη μας τα διαφορετικά και διάφορα συμφέροντα, αλλά κυρίως ερωτώ ποιες είναι οι σχέσεις μας με τρίτες χώρες ως προς αυτό. Κύριε Επίτροπε, Κοιτάξτε, καταρχήν, καταρχήν είτε πρόκειται για τα κράτη-μέλη είτε μέσω της Ένωσης καθεαυτής, πρέπει να καταλήξουμε στην εφαρμογή των, υψηλωτά, των, των υψηλωτέρων δυνατών προτύπων δεν μπορούμε να έχουμε πολύ υψηλά πρότυπα στη Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι στην Ορβηγία. μπορούμε. Και επαναλαμβάνω τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την ασφάλεια των επιχειρήσεων, για τα επίγοντα προγράμματα, για την επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτά είναι τα θέματα που θέλουμε δεσμευτικά καν να εγκριθούν από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και επαφές με τρίτες χώρες για ενεργειακά θέματα, με τη Λιβύη παραδείγματο χάρη έχουμε επαφές και νομίζω ότι είναι δυνατόν να συνομιλήσουμε και με τις άλλες χώρες εταίρους μας και γειτονικέ όπως τη Ρωσία και άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα πραγματικό διεθνή ρόλο. Αλλιώς αποτυχίες όπως της ΜΠΕ πρέπει να ξέρουμε ότι οφείλονται στο ότι αυτοί εφάρμοσαν τελείως δικά τους πρότυπα για τις γεωτρήσεις και αν θέλουν να εφαρμόσουν τα πρότυπά τους αυτά και στα χωρικά ύδατα της Ένωσης τότε πρέπει και εμείς να μπορούμε να επιβάλλουμε πρότυπα το ίδιο αυστηρά και με το ίδιο κόστος και για τις γεωτρήσεις στη Λιβύη ας πούμε. Και όχι να δεχτούμε να, γίνει, να συμβεί κάποιο dumping εδώ ως προς το κόστος και την ασφάλεια. Τα πρότυπα που ισχύουν για την Ευρώπη μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού και πρέπει να εφαρμοστούν και αλλού. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις που ήταν διεξοδικές. Και ζητώ συγγνώμη για του τι ερωτησει ερωτήσει 28-32 που δεν θα μπορέσουν να ακούσουν τι απαντήσει παρά μόνο θα τι λάβουν γραπτό. Αλλά δυστυχώ μα πιέζει ο χρόνο σήμερα το απόγευμα και είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε σε ερωτήσει προ την κυρία Γκόγκαν Κουίν. Θα αρχίσουμε με την ερώτηση 33 του κυρίου Τσουκαλά. um, once the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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε φέτος μια ανακοίνωση για την βελτίωση, ε, για την απλούστευση της, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Χρηματοδότησης Έρευνα και πρότεινε σταδιακέ βελτιώσει, αλλά και ρηξικέλευτε αλλαγέ, απαιτώντα την αναθεώρηση τη νομική βάση για την Ευρωπαϊκή Έρευνα και την ε, επανασυρώπηση του θέματο μεταξύ ανάληψη κινδύνων και αποτροπή η ε, πρόληψη. Είχαμε συζητήσει και με τα άλλα κοινωτικά θεσμικά όργανα και με του ενδιαφερόμενου και χρησιμοποιούμε κατά αποκοπή ποσά για τα διάφορα προγράμματα. Έτσι δεν υπάρχει πια υποχρέωση για λεπτομεριακή ανάλυση του κόστους, μια και έχουμε κατά αποκοπή ποσό και συνδέουμε την καταβολή αυτού με τις επιστημονικές εξελίξεις. Αυτή βέβαια η προσέγγιση έχει κάποιες αδυναμίες, γιατί είναι χρονοβόρες οι διαπραγματευτικές διαδικασίες και επίσης ε, εξαρτάται και από τους ενδιαφερόμενους η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώ όλες τις συνέπειε αυτή τη διαδικασία πριν υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσει. Πάντω για το 7ο ερευνητικό πλαίσιο, ο μέσος ε, τρόπο, ο μέσο τροπο ο μεσος η προθεσμία είναι 340 μέρε. Συντομότερο από το προηγούμενο πρόγραμμα, το έκτο. Βέβαια μπορούμε να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τι διάφορε διαδικασίε. πάντως η συγκριτική αξιολόγηση δείχνουν ότι ε, η μονοετής αυτή προθεσμία δεν είναι πολύ αργή για σημαντικά και μεγάλα επίβολα προγράμματα. Χρειάζεται να επιτύχουμε και μία εναρμόνιση των εθνικών επιδετικών προγραμμάτων για την έρευνα. Βέβαια, τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα συνέβαλαν στο στόχο αυτό και σίγουρα οι κοινέ πρωτοβουλίε ε, θα καταλήξουν σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει πρόσφατα και δυνατότητα για εξωτερική χρηματοδότηση. Και μάλιστα ε, high risk και high gain προγράμματα αναμένονται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Βέβαια, προκαταρκτικές αναλύσει έδειξαν ότι η διαδικασία επιλογή του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου είναι επιτυχής για τέτοιου είδου προγράμματα υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδου. Και μάλιστα οι δράσει ε, Marie Curie θα μπορέσουν να ανατρέψουν ε, την ισχύουσα τάση για διαρροή εγκεφάλων. Από το 1994 οι δράσει Marie Curie επέτρεψαν την ε, δημιουργία πολλών ερευνητικών θέσεων στην Ευρώπη με πολύ ελκυστικού μισθού και με συνολικό προπολογισμό 4,5 δισεκατομμύρια στο 7ο ερευνητικό πρέξιο θα θα ε, επιτρέψουμε σε 50.000 ερευνητέ στην ανάλυση δράσεων και θα βελτιώσουμε και τη σύμπραξη μεταξύ ε, ιδιωτικού και κρατικού τομέα, προκειμένου να ετοιμαστούν οι ερευνητέ για την ένταξή του στην αγορά εργασία. Οι δράσει Marie Curie έχουν ε, απλουστευθεί με μια ενιαία υποτροφία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα το θέμα τη διαρροή διαφυγή εγκεφάλων. Σα ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε. Ο κύριο Τσουκαλά θα υποβάλει την πρώτη συμπληρωματική, μετά ο κύριο Ρούμπιχ και κατόπιν η κυρία Τσικάου. Για μισό λεπτό κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την απάντησή της. Η ερώτηση που υπέβαλα στόχο είχε να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η Ευρώπη παρόλα τα υψηλόφρονα και υψηπετή της σχέδια εξακολουθεί να καθυστερεί σε σχέση με τους στόχους της Λισαβόνας έτσι όπως αυτοί τέθηκαν από την αρχή με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού να έχουν 30% μερίδιο στην βιβλιομετρική αγορά, την Αμερική με 28% και την Ευρώπη πίσω. Ίσως η ύψιστη ποιότητα που ζήτησε για τα μέτρα για τις βυθομετρήσεις ο κύριος Έτιγκερ να, πρέπει να ισχύσουν και για την έρευνα. Ευχαριστώ. Thank you sehr geehrte äh, κυρία Επίτροπε, ε, αυτή τη στιγμή στην έρευνα λαμβάνει χώρα μια πολύ έντονη έρευνα με το πρόγραμμα ΙΤΡΕ. Οι περικοπές ε, αυτή τη στιγμή συζητούνται ε, ευρέως και το Κοινοβούλιο εδώ απορρίπτει αυτό το πλαίσιο σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα αναδιαπραγματευτεί για το ΙΤΡΕ. Κύριε Τσικάο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, το ερώτημά μου σχετίζεται με το ποσοστό χρηματοδότησης που δίνουμε στην έρευνα, ειδικά όμως για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτηθούν για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά πρότυπα χρηματοδότησης, ώστε και τα πανεπιστήμια να, να πάνε υπόψη το κριτήριο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους βουλευτές που έθεσαν αυτά τα ερωτήματα. Εξάλλου το τελευταίο αυτό θα το θέσουμε και σε δύο ακόμη ερωτήματα που σχετίζονται με αυτό. Πρέπει να τονίσω ότι χρειάζεται μια διαθεσμική συμφωνία για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή Ήτρε και την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού στο Κοινοβούλιο αλλά και με το Ελεκτικό Συνέδριο ώστε να υπάρξει επιτέλους μια κοινή πολιτική για αυτό τα σημαντικά θέματα. Οι κανόνες που διέπουν ή που θα διέπουν στο μέλλον τα, προγράμματα, τα ερευνητικά προγράμματα πρέπει να είναι βέβαια συνεπείς μεταξύ τους και όσοι ζητούν ε, χρηματοδότηση για αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, είτε είναι ερευνητικά κέντρα, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε εταιρείε, πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πώ εφαρμόζονται οι χρηματοδοτήσει τη Ένωση. Δέχομαι λοιπόν απόλυτα ότι είναι λογική η ερώτηση αυτή και γι' αυτό και εμείς έχουμε ζητήσει απλοποίηση πρόγραμμα το οποίο συζητούμε ακόμη γιατί συνειδητοποιούμε και εμείς ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών γιατί η απλοποίηση είναι προτεραιότητα κλειδί για ολόκληρη την Κομισιόν και πρέπει να υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος τρόπος που να τον γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Για το θέμα της ΙΤΕΡ και η προηγούμενη θητεία και αυτή, και, και αυτή της Κομισιόν αναγνώρισαν ότι χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη και συνεπής απάντηση αλλά δεν έχει λήξει η συζήτηση του θέματος. Ξέρω ότι και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για το από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα αλλά θεωρούμε ότι γενικά μπορούμε να έχουμε τεράστια ωφέλη από μια επιτυχή τέτοια πολιτική γιατί δεν αφορά καθαρά και μόνο την κοινότητα, την ένωση αλλά έχουμε και διεθνείς εταίρους ως προς αυτό το θέμα και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με αυτούς για να μπορέσουμε το πρόγραμμα να το προωθήσουμε με τη συνεργασία σας και την στήριξή σας φυσικά. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Όπως είπα και από την αρχή μας λείπει αρκετός χρόνος και πρέπει στις 8 και 4 να περάσουμε στις ερωτήσεις προς τον κύριο Χάρμ. Γι' αυτό φοβάμαι κύριε Κέλλη ότι δεν θα προλάβετε. Ούτε τις 37, 38 και 39 και 40 και 41. Επόμενο ερώτημα λοιπόν του κυρίου Παπα-Νικολάου το 34. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η στρατηγική 2020 στοχεύει σε βιώσιμη ανάπτυξη και το Αναπτυξιακό Συμβούλιο το έχει αναγνωρίσει. Προφανώς η λεγόμενη smart growth σημαίνει καινοτομία και έρευνα. Πρέπει λοιπόν να ενδυναμωθούν όλοι οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας και το κλειδί για τη μελλοντική ευμερία της Ένωσης βασίζεται στις ιδέες που θα έχει έτσι ώστε να υποφεληθεί ο κόσμος ολόκληρος. Για να υπάρξει λοιπόν μια καινοτόμα ένωση πρέπει καταρχάς να ενδυναμώσουμε την αριστεία και τη γνώση που έχουμε για τα δεδομένα που αφορούν το θέμα αυτό. Υπάρχει υπάρξει διεθνής αναγνώριση της Ευρώπης ως προς αυτό και αυτό αναγνωρίστηκε τον Ιούλιο του 2009 από μια επιτροπή έξι εμπειρογνωμόνων διεθνή. Βέβαια δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί κανένα πρόγραμμα αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε αποτελέσματα ας πούμε στο Λονδίνο έχουν υπάρξει θεαματικά αποτελέσματα για την ε, μεταμόσχευση οστών με τη χρησιμοποίηση βιοδραστικών ε, συστατικών και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία. Επίσης έχουν υπάρξει αποτελέσματα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος με τη βοήθεια της γενετικής κάτι που θα βοηθούσε ιδιαίτερα τους καρδιοπαθείς. Επομένως υπάρχουν σχέδια που μπορούν να γεννήσουν τελείως καινούργιες ιδέες καινοτόμε και να βοηθήσουν την κοινωνία ολόκληρη. Και τέλος, έχουμε πετύχει επίσης να στηρίξουμε εθνικά ερευνητικά προγράμματα σε πολλές χώρες όπως τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία καθορίζοντας διεθνή πρότυπα αριστείας και με την καταλληλότερη χρήση των ε, κονδυλίων που διαθέτουμε για την έρευνα μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη πρωτοπόρο. Ευχαριστούμε ο κύριος Παπα-Νικολάου για συμπληρωματική. Πράγματι η έρευνα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καινοτομία και η καινοτομία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Θα ήθελα σε συνέχεια των όσων μας είπατε να ρωτήσω το εξής. Μας αναφέρατε το Λονδίνο, μας αναφέρατε την Πολωνία, την Σουηδία αν θυμάμαι καλά, μας αναφέρατε την Πορτογαλία μόνο από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Έχουμε περισσότερα στοιχεία ιδίω για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε σχέση με καλές νέες ιδέες, σε σχέση με απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων προς την στόχευση την ερευνητική ε, δίνουμε έμφαση με δεδομένο ότι οι χώρε αυτέ έχουν πολύ χαμηλού δείκτε στην ανάπτυξη και αναφέρομαι βεβαίω στην ελλάδα αναφέρομαι στην ισπανία και σε άλλε χώρε του ευρωπαϊκού νότου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, δυστυχώς δεν έχω συγκεκριμένε πληροφορίε για τι χώρε του Νότου. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο στηρίζει τις απαντήσεις του σε θέματα αριστείας, άσχετα με τη χώρα, άσχετα με το ερευνητικό κέντρο που υποβάλλει το αίτημα. Δεν λαμβάνει υπόψη τέτοιου κριτήρια, παρά μόνο την αξιοκρατία και την αριστεία σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Γι' αυτό μάλιστα έχει αποκτήσει τέτοια έγκλη διεθνώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, γιατί έχει αναγνωριστεί η αξιοκρατική του προσέγγιση και η στήριξη των αποφάσεών του μόνο σε θέματα αριστείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα θα πρέπει να συνεχίσει περαιτέρω την συνεργασία του με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μάλιστα του χρόνου θα υποβάλει μια νέα δυνατότητα ε, χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης σε προκαταρκτικές φάσεις της ε, καινοτομίας. Στην επαλήθευση, για παράδειγμα, ενός εμπορικού σχεδίου μέσω προτύπων δοκιμών, πιστοποίηση αγοράση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα άξιο πνευματικής προστασίας δικαίωμα. Νομίζω ότι μπορούμε να θαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει καταλήτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι πολλές χώρες και του Νότου εξετάζουν αυτό το, το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας υπό το πρίσμα της ε, ανάγκης θέσπισης αντίστοιχων συμβουλίων και στη, στο εσωτερικό τους. Είναι παράδειγμα προς αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας. Περνούμε στην ερώτηση 35 του Πάτε Κόμπ Κάλαχερ για τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αυξήσει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις βοηθήσει να φέρουν τους καρπούς καινοτομία τους στην αγορά. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει τα ερευνητικά προγράμματα προσιτά στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, απλουστεύοντα το μέτρο του δυνατού τη διαδικασία και εξασφαλίζοντα τη χρηστή ε, δημοσιονομική διαχείριση. Από αυτή την άποψη μειώσαμε την ανάγκη των πιστοποιητικών ελέγχου, ε, τους ελέγχους ε, εξάντε για την χρηματοπιστωτική δυνατότητα, αλλά χρειάζονται φυσικά περισσότερες απλουστεύσεις και προσπάθειες. Εκδώσαμε την ανακοίνωση περί που επίσημα δώσαμε στο Συμβούλιο στις 29 Απριλίου και στο Κοινοβούλιο. Βέβαια προτείνονται και μέσο και μακροπρόθεσμα μέτρα όπως ε, κατά πληρωμές για να καλυφθεί το διαχειριστικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα ερευνητικά προγράμματα και θα προτείνουμε αλλαγές και στο νομικό πλαίσιο αν παραστεί ανάγκη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τελευταιο έβδομο ερευνητικό, πρόγραμμα πλαίσιο κάποια ειδικά προγράμματα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ειδικού προπολογισμού για αυτές. Το 14,7% πέρασε ε, στο 15,7% για τα προγράμματα συνεργασίας. Ξεπεράσαμε λοιπόν τον στόχο του 15% στην ε, νομοθεσία πλαίσιο. Φυσικά θα παρακολουθούμε εκ του και στην πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Και τα Eurostars ε, είναι ένα πρόγραμμα κοινό μαζί με το Eurek, το Εύρικα που φέρνει, κοντά, φέρνει στη συνεργασία 26 χώρε μέλη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν προγράμματα που θα είναι κοντά στην αγορά. Αλλά και το δίκτυο επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 2008 προσφέρει υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Φυσικά όλα αυτά γίνονται σε πλήρη συμπληρωματικότητα με τα εθνικά σημεία επαφής που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν καλύτερα για τις δυνατότητες ε, του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, για τις ε, εταιρικέ σχέσεις, τις συμπράξεις, τις κοινέ δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συμπερίληψη των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν στα ερευνητικά προγράμματα. Μέσω των μέτρων αυτών περιμένουμε ότι 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν από το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Τέλος, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης, ειδική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τεθεί στο διαδίκτυο το 2011. Έτσι θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράμματα και με ειδικέ πληροφορίες και online ε, κατάρτιση θα βελτιωθούν οι δυνατότητες τους για αξιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Καλώς. Ερώτηση του κυρίου Γκάλαχερ και του κυρίου Κέλλη συμπληρωματική γιατί δυστυχώς ε, τη δική του ερώτηση θα προλάβουμε να την απαντήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις ε, διεξοδικές της απαντήσεις. Και να πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, κέρδιας και νευραλικής σημασίας για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ραχοκοκαλιά ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή τους στην οικονομική ανάκαμψη θα είναι σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την ε, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην καρδιά του προγράμματός της. Θα πρέπει όμως να αυξήσουμε το επίπεδο συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γκέογκαν Κουίν, την Επίτροπο, τι πρόκειται να κάνει για να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιλήσουν χρηματοδότηση από τα ερευνητικά προγράμματα που εμπίπτουν στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Ο κύριος Κρόλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την απάντηση του, της Επιτρόπου. Να πω το εξή. Το 90% των νέων προϊόντων που προέρχονται από προγράμματα προσανατολισμένα στην έρευνα ε, προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές αφορά στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων και της ε, προστασίας τους. Υπάρχουν λοιπόν άραγε στην ε, Επιτροπή κάποια σχέδια για να έχουμε την προστασία των δικαιωμάτων αυτών και ε, υπάρχουν ίσως και νέες δυνατότητες για την έρευνα. Ο κύριος Κέλλη. Πρώτα απ' όλα ε, πιστεύω ότι ε, όσον αφορά τα αποτελέσματα της δουλειάς που κάνετε Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται αυτή ε, στους ανθρώπους ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα γίνουν ακόμα πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Η Επίτροπος. Κοιτάξτε, χαίρομαι πάρα πολύ ε, που μου δώσατε τη δυνατότητα να απαντήσω και εγώ στη μητρική μου γλώσσα Ελπίζουμε ότι οι έρευνες που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009 θα βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την ε, ταχύτητα της ε, διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και με τα προγράμματα που προβλέπονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, υπάρχουν νέες αποφάσεις ε, για συνεργασία για το 2011 και οι αποφάσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς ε, σε μεγαλύτερη συνεργασία. Εμείς ε, θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, ε, τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν το 2012 και το 2013. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά τον κανονισμό ε, πριν από λίγο αναφέρθηκα ότι μας ενδιαφέρει και η απλούστευση. Ορισμένα πράγματα μπορούν να εφαρμοστούν ε, αμελητή στο πλαίσιο του ε, προγράμματος που, και του πλαισίου που ισχύει. Οι δομές μπορούν να βελτιωθούν με διάφορους τρόπους. Η ίδια η Επιτροπή ερευνά και μικρές αλλαγές ε, στο ρόλο της ε, Κομισιόν έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό το μέσο κόστος. Και ίσως αναθεωρηθούν και οι κανονισμοί που αφορούν ε, στον, στα λογιστικά. Δίκιο έχετε όταν μιλάτε για τα νέα αυτά προγράμματα Όλα αυτά τα προγράμματα προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν δύσκολο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, αλλά μία από αυτές είναι αυτή που είπατε, τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ ε, προεδρεύω στη ομάδα τη Επιτροπή ε, για την Καινοτομία και ένα από του συναδέλφου μου είναι ο επίτροπο κύριος Μπαρνιέ που ασχολείται ακριβώ με αυτόν τον τομέα. Συνεργαστήκαμε λοιπόν στενά και όταν θα ε, χαραχθεί και θα δημοσιευθεί η πολιτική καινοτομιών στι αρχέ Οκτωβρίου θα δείτε ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει και άλλοι και όπως είπα και εσείς έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, τώρα, ε, όσον αφορά ε, τα δεδομένα που αποθηκεύονται και υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, ε, ιδιωτικές εταιρείες που θεωρούν ότι υπάρχει ένας χώρος για αυτές τις ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευθούν. Εμείς θα θέλαμε όταν θα δημοσιευθεί ε, το βιβλίο μας ε, για τις καινοτομίες αυτό να εκλειφθεί ως μια σοβαρή προσπάθεια ε, εκ μέρους Κομισιόν να καταθέσει τολμηρές προτάσεις που βεβαίως και πρέπει να συζητηθούν τολμηρές προτάσεις που εξετάζουν αυτά τα προβλήματα και τα ε, προσκόμματα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι εταιρείε που ενδιαφέρονται σε τέτοιου είδου ε, θέματα θα κατανοήσουν ότι η Κομισιόν είναι πρόθυμη να απαντήσει ε, θετικά και χρειαζόμαστε υποστηρικτές. Ο κύριος Κέλλη είπε ότι ο... όποιος προλάβει πιο γρήγορα κερδίζει σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα. Αυτό αφορά τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς, ε, την πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το... τα venture capital που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα ερευνητικά έργα, τα ερευνητικά κέντρα, συγγνώμη, τα πανεπιστήμια, οι ιδιωτικές ε, και κρατικές επιχειρήσεις, αλλά και στο Κοινοβούλιο όταν εξετάσαμε όλα αυτά τα θέματα για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη νέα πολιτική περιλήφθηκαν στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το διαπιστώσετε όταν δημοσιευθεί η νέα πολιτική με τις προτεραιότητες. Φυσικά θα πρέπει να προκολουθήσουμε την εφαρμογή της διαδικασίας, να την στηρίξουμε και να εξασφαλίσουμε και συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Πολύ διεξοδικές οι απαντήσεις και χρήσιμες. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις προς τον κύριο Χάν και λυπούμε για όσους κατέθεσαν τις ερωτήσεις 36 έως 41 γιατί δεν προλάβαμε να τις απαντήσουμε. Θα τις λάβουν γραπτός λοιπόν τις απαντήσεις. Μας πιέζει ο χρόνος γιατί οφείλουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 8.30. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση παριθμό 42 του κυρίου Πόσελτ στρατηγική για το Δούναβι και ευρωπεριοχές. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα τέταρτο να διεκπεράσουμε και τις τρεις ερωτήσεις, ένα πεντάλεπτο για την καθεμία δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα που έχει τεθεί η προοπτική συνεργασίας ανάμεσα στη Βαβαρία και την Αυστρία και την Τσεχία πράγματι ε, αυτή είναι μια θαυμάσια προοπτική για μια περιοχή η οποία αφορά 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Ενδιαφέρει η εξέλιξη της περιοχής σε πολιτιστικό, τουριστικό επίπεδο αυτή η διάσταση νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και σε σχέση με τη στρατηγική του Δούναβη. Ο τομέας αυτός ε, έχει τεθεί στις διάφορες διαβουλεύσεις κυρίως ε, όσον αφορά στον τουρισμό η περιοχή αυτή ε, έχει λάβει ιδιαίτερη προσλάβει ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο της ε, πολιτιστικής ε, συνεργασίας έχουν κατεθεί πολύ ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις, κυρίως όσον αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο. Τώρα, ως προς την προώθηση αυτών των περιοχών, η Τσεχία, η Αυστρία και η Βαβαρία σε αυτές τις χώρες εφαρμόζονται διάφορα προγράμματα συνεργασίας ύψους ε, περίπου 430 εκατομμυρίων ευρώ για την τρέχουσα περίοδο. Νομίζω ότι το ποσό είναι αρκετά ενδιαφέρον και να πόκειται πλέον στις ε, ενδιαφερόμενες αυτές περιοχές ε, να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες στο μέγιστο. Η ιδέα του να υπάρχει μία διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό για μένα είναι αποτελεί μια θαυμάσια ιδέα και θα οδηγήσει και στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής. Ο κύριος Πόσελ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πίτροπε για την πολύ καλή σας απάντηση. Εν τω μεταξύ έχει εμφανιστεί ε, κάτι καινούριο το Φίλσεν φαίνεται το 2015 η ε, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί η πολιτιστική συνεργασία στην ε, Ευρωζώνη. Κατά πόσο αυτό θεωρείται ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Ε, προφανώς εγώ είμαι 100% πεπισμένος ότι ειδικά ως προς την πολιτισμική συνεργασία η διασυνοριακή συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη, διότι ε, το πολιτιστικό πλαίσιο είναι διασυνοριακό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πολιτισμικό στοιχείο να είναι ένα καθοριστικό στοιχείο ε, της συνεργασίας ε, και αυτών των περιοχών στο Δούναβι. Με την πολιτισμική ε, πρωτεύουσα το Πίλσνερ προφανώς ε, θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ε, κίνημα. Thank you, Commissioner. Thank you, Πάμε στην ερώτηση παριθμών 43 του κυρίου Κρόουλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω ότι πριν από λίγες μόνο ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε θετικά Προτείνει λοιπόν εδώ την ε, οικονομική ενίσχυση που ε, υπερβαίνει κατά τη τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια πρόταση και γνωρίζετε ότι για να υλοποιηθεί η πρόταση πρέπει να δοθεί και η έγκριση από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο. Και θα ήθελα σύντομα να σας υπενθυμίσω περί τίνος πρόκειται. Στις 19 Νοεμβρίου του 2009 εντοπίστηκαν οι πρώτες ζημιές, καταγγέλθηκαν οι πρώτες ζημιές και η αίτηση κατατέθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2010, την τελευταία ακριβώς ε, προθεσμία που ήταν περίπου 10 εβδομάδες, την τελευταία ημέρα. Μετά χρειάστηκε να υπάρχουν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Στις 24 Μαρτίου εμείς ε, στείλαμε ένα ερώτημα προς τις Ιρλανδικές Αρχές. Μας απαντήθηκε γύρω στα μέσα Ιουνίου και το πρόβλημα είναι ότι λόγω ε, του, συνόλου της διαπιστωμένης ζημιάς δεν επιτυγχάνεται το κατώτατο όριο αναγνώρισης εθνικής καταστροφής. Άρα δηλαδή πάμε σε άλλη κατηγορία. Κατά πόσον η ζημιά αυτή θα μπορούσε να ε, ταξινομηθεί ως ε, περιφερειακή ζημιά. Και για να γίνει όμως κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνουν έρευνες και αξιολογήσεις. Έγιναν όλα αυτά. Τώρα πλέον έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Στις 14 ε, Σεπτεμβρίου καταθέσαμε την πρότασή μας με βάση την οποία για να καλυφθούν οι δαπάνες του δημοσίου που προέκυψαν λόγω αυτής της ε, καταστροφής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει το απαραίτητο ποσό που όπως σας είπα ξεπερνάει κατά τα 13 εκατομμύρια ευρώ ε, υπό την αίρεση της έγκρισης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο σύντομες συμπληρωματικές, το πολύ μισό λεπτό. Κρόλι και Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για τις απαντήσεις του και να πω ότι μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι ότι προσθέτει συνέχεια έξοδα στην αρχική κοστολόγηση, αποτίμηση των ε, ζημιών. Και μάλιστα στη δική μου γενέτειρα που ε, έχουμε μόνο 5.000 ανθρώπους, 19 επιχειρήσει ε, εξακολουθούν να παραμένουν κλειστέ εξαιτία των ζημιών που υπέστησαν από τι πλημμύρε. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και πιο μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείριση και να μην περιοριστούμε μόνο στην άμεση απάλυση των ε, ζημιών. Ο κύριο Κέλλη και μετά ο κύριο Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για τις απαντήσεις και για τη χρηματοδότηση, παρόλο που δεν φτάσαμε στο εθνικό κατόφλι έχετε σκοπό να τροποποιήσετε τα κριτήρια για το εθνικό κατόφλι. Γιατί το να ισχύουν τέτοια κριτήρια για όλε τι χώρε, ε, αποβαίνει βάρος των μικρό χωρών και εξαρτάται και από την θεομηνία. Ε, πολλές φορές θα αφαιρεθούν σε δυσμενέστερη θέση οι μικρότερε χώρε από τι ε, μεγαλύτερε. Ο κύριο Γκάλαχερ, θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του υπαλλήλου τη που συνεργάστηκαν στενά με τις αρμόδιες αρχές στην Ιρλανδία. Και όπως είπατε, η άμεση αντιδράση εκτιμήθηκε ιδιαίτερος και τα 30 εκατομμύρια που δόθηκαν αρχικά. Μήπως θα μπορούσατε όμως να συστήσετε στους συναδέλφους σας μια τροποποίηση του κατοφλίου, γιατί το κατόφλι για την Ιρλανδία ήταν περίπου ένα δις και φυσικά δεν φτάσαμε σε αυτό το κατόφλι. Ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τα καλά σε αυτά λόγια ε, θα τα διαβιβάσω περαιτέρω στους ε, συνεργάτες μου οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Όσον αφορά στους ε, κανόνες για το Ταμείο Λεγγύης, οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ότι το κατώτατο όριο πρέπει να είναι 0,6% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η κατώτατη, το κατώτατο ποσό που σημαίνει στην περίπτωση της Ιρλανδίας 935 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να είναι τουλάχιστον η ζημιά. 3,5 δις είναι το ανώτατο όριο. Αυτό βέβαια αφορά 3-4 μεγάλα ε, ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία ε, κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους λόγους γιατί η Κομισιόν ήδη το 2005 προέβη σε προσαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός, απλουστεύοντας το κατώτατο όριο, έτσι ώστε να υπάρχει μείωση του κατώτατου ορίου για μεμονωμένα κράτη-μέλη. Από την άλλη βέβαια να υπάρχει και διασύνδεση των ε, δύο κατηγοριών που αφορούν στις εθνικές και στις περιφερειακές καταστροφές. Δεν θέλω να σας κρύψω ότι για την αποζημίωση δαπανών έχουμε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων από αυτές που μπορούμε να εικονοποιήσουμε. Και αυτό όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αξιολογήσεις που κάνει δεν καταλήγει στο ότι πρέπει να υπάρξει αποζημίωση. Στόχος μας λοιπόν είναι να επιταχυνθεί βέβαια η διαδικασία αλλά να υπάρχουν και ε, κάποια νέα κριτήρια. Γιατί όπως βλέπετε στην περίπτωση της πατρίδας σας, της Ιρλανδίας, ε, μιλάμε για δέκα περίπου μήνες. Ε, αν προσθέσουμε και κάποιες άλλες μέρες θα φτάσουμε μέχρι τον ένα χρόνο μέχρι να εκταμιευθεί τελικά το ποσό. Και κάτι άλλο που σας είπα, τα κριτήρια, το τι μπορεί να χαρακτηριστεί καταστροφή αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Λεγγύης μπορεί να καλύψει μόνο θεομηνίες. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καλύπτονται και άλλου είδους καταστροφές. Παραδείγματος χάρη ε, καταστροφές που οφείλονται στην τεχνολογία. Έγινε μάλιστα αυτή η σχετική πρόταση το 2005 και απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν πολλές καταστροφές, εγώ προετοιμάζω μία προσαρμοσμένη πρόταση, η οποία λαμβάνει υπόψη της την εμπειρία των τελευταίων ετών. Ελπίζω λοιπόν ότι τώρα πλέον ορισμένα κράτη τα οποία τους τελευταίους μήνες έτυχαν της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ελπίζω τα κράτη αυτά να προσαρμοστούν και στο μέλλον να έχουμε ένα ταμείο λεγγύης το οποίο θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα πολύ γρήγορα θα περάσουμε στο ερώτημα του κ. Χάρν. Αλλά και εσείς πολύ σύντομα κύριε Επίτροπε, πολύ σύντομα. Γιατί η προηγούμενη απάντηση ήταν μακροσκελής. Και σε δύο λεπτά πρέπει να κλείνουμε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, η νέα Βρετανική κυβέρνηση ε, έχει δεσμευθεί για, σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τοπική κοινωνία. Ακόμα δεν είναι απόλυτα σαφές πώς θα διαμορφωθούν οι νέες δομές. Κατόπιν τούτου και εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ αμετάκλητα. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, θα δούμε πώς θα ε, διαμορφωθούν οι νέες δομές, ε, οι νέες αρχές διαχείρισης, θα υπάρξει και η σχετική προσαρμογή των προγραμμάτων. Ελπίζω βέβαια, παρότι οφείλω να ομολογήσω ότι ανησυχώ, ελπίζω να μην προκύψει υπερβολική καθυστέρηση στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Ο κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος για να σεβαστώ τον χρόνο μας. Κύριε Επίτροπε, εγώ είχα ρωτήσει στο ερώτημά μου τι διαβουλεύσεις έχουν ήδη γίνει μεταξύ Κομισιών και Κυβέρνησης του ΙΤΑΒ. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει γίνει καμία διαβούλευση. Δεν μου απαντήσατε. Και μπορείτε να μας πείτε σήμερα αν τα κριτήρια και της προσθετικότητας και της ε, ουδετερότητας θα γίνουν σεβαστά. Η επάνηση είναι απλή. Ε, δεν έχει υπάρξει ανάληψη επαφών και η ιδέα της ε, βραχυπρόθεσμης ε, χρηματοδότησης πρέπει να ισχύει και στο μέλλον, αν αυτό εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ για την καθαρότατη αυτή απάντηση. Λίγη εδώ η ώρα των ερωτήσεων και θα επαναλάβουμε στα σενέα.